προτείνει την, ε, τον έλεγχο τη εντολή του κυρίου Ζακ Κολομπιέ και προτείνει την έγκριση τη θητεία του από τι 2 Φεβρουαρίου 2018. Υπάρχουν παρατηρήσει. Ωραία. Εγκρίνεται λοιπόν ε, η εντολή.